Συνάδελφοι, λέει κυρία Χιούμπνερ, πολλέ πίσει έχουν αργήσει, αλλά μην αργήσει η συνεδρίασή μα. Δεν έχω έτσι καλώ ιδέα τι ώρα μπορεί να έρθουν οι συνάδελφοι. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κανένα πέντε λεπτάκια ακόμα, αλλά από ό,τι ακούμε Υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις πτήσεις στην Ευρώπη. Άρα δεν θα έρθουν και πολλοί συνάδελφοι. Άρα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι όσοι να δείτε στο ίντερνετ τη συνεδρίασή μας και επίσης σας ενημερώνω ότι έχετε λάβει ε, στις 20 Φεβρουαρίου του 2018 ε, το σχέδιο της ε, ημερησής διατάξεως και στο μεταξύ όμω συνέβησαν τα εξή τρία. Πρώτα πρώτα ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ απεφάσισε να επανέλθει στην ε, ομάδα εργασία σε σχέση με την πρότασή του γιατί είχε ζητηθεί από τον πρώτο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκθεσή του να αναβληθεί. Άρα σήμερα δεν τον έχουμε εδώ. Επίσης, δεύτερο θέμα, επειδή είχε κάποια προβλήματα η νομική επιτροπή όσον αφορά την παρουσία συναδέλφων για την έκθεση που αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία της Διοργανικής Συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία ζήτησαν να αναβληθεί η κοινή συνεδρίαση των δυο μας επιτροπών. Και τρίτον, κατά το οποίο είναι μια λέξη τελευταία στιγμή. Ο George Σέπφλιν, ο εισηγητής του ECR, θα έρθει, αλλά αργότερα. Γιατί έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να περαστεί από την αρχή της συνεδριασής μας. Οπότε είπαμε ότι θα τον περιμένουμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Και ο κ. Βοητσόφσκι ελπίζουμε να έρθει επίσης. Επίσης εκ μέρους του Βίλανδη η Mercedes θα μας ε, ενημερώσει. Τέλος πάντων αυτά μόλις αρχίσει το κυρίως πιάτο της συνεδρίασης. Οπότε αν δεν έχετε κάποια ένσταση για αυτές τις αλλαγές στη μέση διάταξη, τότε θεωρώ ότι την εγκρίνετε με αυτές τις τροποποιήσεις που σας ανέφερα και πάμε στο σημείο 2 αυτής, που είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου να σας πω τα σχετικά με το Brexit αύριο, γιατί έχουμε σημείο για το Brexit. Σήμερα όμως να σας ενημερώσω για το εξής. Η συνάντησή μου με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας της Βιέννης των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήρθε ο Μάικλ να με βρει για να δούμε τι δυνατότητες στενότητες συνεργασίας υπάρχουν μεταξύ εκείνων και ημών. Και όπως θα θυμάτε, θα θυμάστε, είπαμε ότι δεν θα είναι εδώ τότε η Μπάρμπαρα Σπινεριτή γιατί την έκθεσή της που αφορά την υλοποίηση του χάρτη ανθρωπινών δικαιωμάτων. Οπότε θα μπορούσαμε με την ευκαιρία που θα δούμε τον Διευθυντή να αξιοποιήσουμε καλύτερα την έκθεσή σου, Μπάρμπαρα. Μέχρι τώρα συνεργάζονται ε, οι υπηρεσίε υπηρεσίες των δικαιωμάτων με την ΠΕΤΗ και με την employment. Αλλά νομίζω ότι και δύο πλευρές έχουν να κερδίσουν αυτή τη συνεργασία. Οπότε θα κρατήσουμε επαφή και θα δούμε πότε είναι η πιο σωστή στιγμή ο κύριος Ο. να έρθει να μας επισκεφθεί. Τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση όσον αφορά τι προτάσει των συντονιστών. Η συνεδρίαση τη 23η Ιανουαρίου απέφερε τα εξή. Θα ανατεθούν οι εξή ε, γνωμοδοτήσει. Πρώτα-πρώτα. Έχουμε την έκθεση της ΕΝΒΙ για την οποία θα λάβουμε σχέδιο συμβουλευτικής ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και θα τον ελάβουν οι σοσιαλδημοκράτες και συγκεκριμένα με Μπρέσο. Η δεύτερη έκθεση για την οποία πρέπει να γνωμοδοτήσουμε είναι μια έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά ε, την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ορίστηκε εισηγητής ο κύριος Μάσιμο Καστάλτο του EFDD. Τρίτη έκθεση. Η τρίτη γνωμοδότησή μας αφορά έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αυτό το ανέλαβε ο ΕΛΚ και η συγκίτρια θα είναι η υποφαινομένη. Τέταρτον, πάλι για την Οικονομική Επιτροπή. σε σχέση με την θωράκιση της δημοσιονομικής ευθύνης και τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές και κατευθυντήριες για τα κράτη-μέλη. Σοσιαλδημοκράτες. Συγγνώμη, οι σοσιαλδημοκράτες η κυρία Κλόντια Ταπαραντελ. και η τελευταία φορά την ε, Λίμπη όσον αφορά ε, τις παραβιάσεις Τη αρχή του κράτου του δικαίου από την Πολωνία. Αυτό το αναλαμβάνει η κυρία Μάιτε Παγκαθαουρτουντούα για τους φιλελευθέρους. Αλλά τελευταία είναι οι γνωμοδότες για την ΕΚΟΝ όσον αφορά τα απαιτούμενα ε, όσον αφορά επενδυτικές εταιρείε, που είναι κανονισμός του Κοινοβουλίου όμως για αυτή την τελευταία αποφασίσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο. Η κατάσταση στην Ουγγαρία. Η Μάιτε Παγκαθαρδουντούα είναι η εισηγήτρια. στη συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ 1η Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα λίγη προθεσμία των τροπολογιών και ας δώσουμε στην Μάιτε ευθύ αμέσως τον λόγο να μας παρουσιάσει τα θέματα της. Μάλιστα, μάλιστα, έτσι είναι πρόεδρε. Έληξε η προθεσμία ε, για τις τροπολογίες, είχαμε πολλές ε, τροπολογίες, περίπου 32. Βλέπετε επομένω ότι προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή. Οπότε και πολλές από αυτές τις απόψεις κατευθύνονται προς το αυτό. Δηλαδή, έτσι θα προσανατολίσουμε και εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο έργο μας. Τα ξαναείπαμε, δεν είχαμε πάρα, πολύ, πολλά περιθώρια, όπως γνωρίζετε πιεζόμαστε. Ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και ότι θα έπρεπε να είναι ευσύνοπτο το κείμενο, πάντως πολλοί από εμά ανησυχούν θα πρέπει η Ουγγαρία να αναγνωρίσει την Επιτροπή της Βενετίας. Αυτό είναι αντικείμενο κάποιων τροπολογιών και δική μου. Οπότε, είπαμε ότι η ιδιότητα Ευρωπαίου πολίτη δεν είναι μόνο κάτι που έχει να κάνει με το να είναι κανείς από κάποιο κράτος μέλος. Είναι κάτι ευρύτερο. Αυτό θα πρέπει να θίξουμε στην γνωμοδότηση. Και από πολλές πλευρές αμφισβητούν πάρα πολύ σημαντικά δόγματα, αξίες, αρχές. Αλλά θα πρέπει εμείς αυτοί που το κάνουν, το κάνουν λόγω ιδεολογίας, το κάνουν λόγω προέλευσής τους. Μα από την άλλη μεριά δεν του ανάγκασε κανεί να ανήκουν στο κλαμπ, στη λέσχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να ξέρει κανεί να, να, να, να ξέρει κανείς με τον μπαίνει στην λέσχη τι αρχές πρέπει να αναδεχθεί, τι είπα να η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άρα και στην προκειμένου λοιπόν αυτό λέμε στην εκθέσή μας. Θα προσπαθήσω τέλο πάντων να ομαδοποιήσω, να, να, τι τροπολογίε τις τροπολογίες από των αδέλφων και στις συναντήσει που θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε όσο πιο επιμελώς γίνεται τη δουλειά. Ευχαριστώ όσους ήρθαν σήμερα, ευχαριστώ όσους συνέβαλαν τις προτάσεις τους και θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο θετική. Ευχαριστούμε Μάιτε για το ΕΛΚ. Ο Κρίστιαν Νταν Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση που και πιστεύω ότι πραγματικά καλύπτει τα πιο ουσιαστικά σημεία. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα κάποιες πτυχές, όπως την ισορροπία των ε, εξουσιών. Εδώ απειλείται κατά κάποιο τρόπο η δικαστική εξουσία και αυτό θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία των εξουσιών, την οποία πρέπει να επανορθώσουμε. Βλέπουμε επίσης ότι οι προτάσεις από μέρους της Βουδαπέστης για νέα νομοθεσία είναι κάθετα αντίθετες με πολλές από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 πρέπει να το χρησιμοποιούμε όταν υπάρχει παραβίαση, κατάφορη παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να υπάρχει και πολιτική βούληση και τα αποτελεσματικά νομοτικά εργαλεία. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την διαδικασία επί παραβάση επανειλημμένος κατά ενός κράτους μέλους και όταν το κράτος μέλος αυτό διαρκώς απαντά ε, συνεχίζοντας αυτές τις παραβιάσεις δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τις δεχόμαστε και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει κατάφορη παραβίαση αυτών των άρθρων και ιδιαίτερα του Δίου. Είμαστε εδώ μπροστά σε μία σαφή κατάσταση πολλαπλών παραβιάσεων οι οποίες συνεχίζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να αντιδράσουμε, αλλά να είμαστε πολύ μετριοπαθείς. Σκοπός μας δεν είναι να ε, καταδικάσουμε εμείς την ε, Ουγγαρία, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση και ο σεβασμός αυτών των αξιών και βεβαίως η Επιτροπή σαν θεματοφύλακας των συνθήκων καλείται να παρακολουθήσει την ε, τήρηση αυτών των αρχών. Εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε μεροληπτική θέση. Έχουμε πολλά παραδείγματα και με την Ουγγαρία αλλά και με άλλες χώρες, όπως τη δική μου χώρα. Εχθές είδαμε λύπη την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας που ήταν ε, συνάδελφός μας ε, στους σοσιαλιστές, η κυρία Ντετσιλέ, η οποία κατηγόρησε την Άννα Γκόμες η οποία μάλιστα ανήκει και στην ίδια πολιτική ομάδα, ναι. να είναι εχθρός της Ρουμανίας, λέγοντας ότι την ελέγχει ο Σόρος. Αυτό είναι μια απειλή που ακούμε πολλές φορές στα Βαλκάνια. Γιατί, γιατί η Άννα Γκόμες τόλμησε να επικρίνει την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Και αυτό μεταξύ συναδέλφων σοσιαλιστών. Πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες και το διακύβευμα είναι πολύ σοβαρό, πρόκειται για το κράτος δικαίου και πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μην είμαστε αμερόληπτοι γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Κάφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι πραγματικά η γνωμοδότησή της είναι πάρα πολύ καλή. Και όπως είπε και η ίδια, οι τροπολογίες σαφώς και θα πρέπει να συμπληρώσουν, να ενισχύσουν τη δική της γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση αφού τροποποιηθεί και αφού συμπεριληφθούν οι σημαντικές τροπολογίες θα πρέπει να ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία για να έχει δύναμη. Όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Πρέντα. Η συζήτηση για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τους ε, τις βασικές μας αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες συζητήσεις, στην Ολομέλεια, όταν παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά έναν ε, μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σεβασμό της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, έναν μηχανισμό που ξεπερνά τα πολιτικά κόμματα, τις παρατάξεις και πραγματικά έχουμε κατά νου να προστατεύσουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει κάθε φορά που υπάρχει μία παραβίαση αυτών των αρχών, όπως παραδείγματος χάρη κράτους δικαίου, θα πρέπει να το αναφέρουμε και να το καταδικάζουμε πέρα από πολιτικές συμπάθειες ή προσεγγίσεις. Σήμερα τα νέα που μας έρχονται από την Ουγγαρία είναι ανησυχητικά. Όσον αφορά τα επιδόματα που παίρνει η Ουγγαρία, ξέρετε και βλέπετε τους αριθμούς υπάρχουν ε, στις τελευταίες μας εκτιμήσεις και θεωρώ πολύ σημαντικό τα χρήματα που συνεχίζει να παίρνει η Ουγγαρία να επαναυπολογιστούν. Θα πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή να παίξει το ρόλο της. Και θα χαρώ πολύ αν ε, οι τροπολογίες που έχω υποβάλει προς αυτή την κατεύθυνση υποστηριχθούν από τους περισσότερους συναδέλφους. Πιστεύω ότι αυτές οι τροπολογίες καθώς και άλλες που αφορούν ε, την ε, Επιτροπή της Βενετίας, τις συστάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή της Βενετίας και η εμπερογνωμοσύνη της Επιτροπής της Βενετίας η οποία είναι μοναδική σε αυτό το τομέα γιατί όπως ξέρετε με τη διαδικασία της παρακολούθησης μπορεί να μας δώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Ε, προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά τις τροπολογίες με την εισηγήτρια και ευχαριστώ πολύ για τη μέχρι τώρα δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR. Mm. Bardzo krótko, Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. E, ja jestem e, wyczulony na kwestie e, το θέμα της, του να δοθεί απάντηση στα προβλήματα της, του κράτους δικαίου και τα θέματα τα συνταγματικά, οι θέσεις μου είναι γνωστές από τους Πολωνούς συναδέλφους. Εγώ θα ήθελα όμως να προσπαθήσουμε να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε το να κατηγορήσει κανείς μια κυβέρνηση ότι παραβιάζει το κράτος δικαίου δεν είναι κάτι το ανώδυνο. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένες παραβιάσεις οι οποίες αφορούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες του κράτους δικαίου. Σαν παράδειγμα συνοπτικές δικαστικές διαδικασίες, κατηγορία εις βάρος των δικαστηρίων ότι δεν λειτουργούν αντικειμενικά, αμφισβήτηση για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος κτλ. Λοιπόν, η έκθεση θα έλεγα έχει κάποια εκρηκτικά στοιχεία. Λέει ότι στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά στον τομέα του κράτους δικαίου μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή. Εγώ δεν θα συμφωνήσω εδώ. Θεωρώ ότι τα ανώτατα αυτά επίπεδα θα πρέπει πάντα να γίνονται δεκτά και σεβαστά. Δεν μπορεί να υπάρχει κατά το δοκούν εκ νέου διερμηνία, ερμηνεία συγγνώμη, ε, των επιπέδων αυτών. Ε, προέρχομαι από μια χώρα ε, στην οποία θεωρώ ότι γίνεται σεβαστό το συνταγματικό δίκαιο της χώρας και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος για τις προτάσεις της εισηγήτριας. Νομίζω ότι οι αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι επακριβέστερες ή καλό θα είναι αν δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένες να μην τις κάνει καθόλου. Η κυρία Σπινέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαϊτέ για την εξαιρετική της δουλειά. Θα συμφωνήσω με όλα όσα αναφέρει. Νομίζω ότι υπάρχει μια υποσημείωση εδώ, ε, η οποία είναι σημαντική και εκεί θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες σε συνεργασία με τους πρασίνους. Ε, θεωρώ ότι η σημερινή κατάσταση στην Ουγγαρία αντιπροσωπεύει έναν σοβαρότατο κίνδυνο παραβίασης των αξιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της συνθήκης. Αυτό στην ουσία οδηγεί στην εφαρμογή του άρθρου 7. Το λέγω αυτό διότι αυτή τη στιγμή αναφερόμεθα στην προσφυγή ε, για την Πολωνία το άρθρο 7, τότε δεν θα είναι πάρα πολύ σωστό κάτι τέτοιο να μην γίνει για κυβερνήσεις και χώρες, άλλες κυβερνήσεις και άλλες χώρες, οι οποίες επιδεικνύουν τις ίδιες συμπεριφορές. Δεν μπορώ εγώ να δεχθώ μια λογική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Τι άλλο να προσθέσω εδώ. Όπως είπα η γνωμοδότηση της Ροής είναι εξαιρετική. Να γίνει ίσως μία αναφορά στο σημείο 8. Στο σημείο 8 της γνωμοδότησης γίνεται αναφορά σε μία σειρά παραβάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν στην Ουγγαρία. Εδώ θα ήθελα να προσθέσουμε παρακαλώ και τα μέτρα τα σχετικά με τη μετανάστευση, τους ετούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και την ελευθερία του συνέρχεστε επίσης. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω συγκεκριμένη αναφορά και στο νέο νόμο της 13ης Φεβρουαρίου, ένα νόμο εξαιρετικά σκληρό εις βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που φροντίζουν ε, τους πρόσφυγες. Εθνικές και ε, διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση της ΜΑΙΤΕ, η σημασία επίκλησης ε, εναλλακτικών ή παράλληλων μηχανισμών με το άρθρο 7 του οποίου η εφαρμογή παρουσιάζεται δυσχερής. Σαν παράδειγμα, ο μηχανισμός που περιγράφεται στην έκθεση Intvelt για την τήρηση του κράτους δικαίου, του κανόνα, των, των κανόνων του κράτους δικαίου και επίσης και το θέμα της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω εδώ. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αυστηροί οι κανόνες της Κοπενχάγης και θα πρέπει να ισχύσουν με αυστηρό τρόπο και για τις χώρες μέλη της Ένωσης, όχι μόνο για τις νέες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πασκάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω όχι να αντικαταστήσω γιατί ποιο τολμά να αντικαταστήσει τον Κάμπρας ο οποίος είναι στην Καταλωνία αυτή την εβδομάδα και δεν μπορεί να είναι μαζί μας για πολιτικούς λόγους. Να πω εδώ και χαίρομαι που συνεχίζω σε αυτά τα οποία είπε η Μπάρμπαρα την τελευταία φορά διαφωνούσαμε λίγο και μου κάνει εντύπωση που διαφωνούσαμε γιατί συνήθως συμφωνούμε. Τώρα όμως θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την Ρούς για την γνωμοδότησή της. Να πω στην Ρούς ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις της. Είναι σαφές να δείξουμε ακριβώς ότι η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ένα κράτος ε, δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε κυρώσεις εις βάρος των δε και όχι εις βάρος των μεν. Και να πω επίσης ότι ο κύριος Τιέρη Κάμπρας, όπως το προβλέπει και η Λίμπε και όπως το πρότεινε και η Μπάρμπαρα, να προσπαθήσουμε ε, να ολοκληρώσουμε την διαδικασία που ακολουθούμε και να ζητήσουμε παρακαλώ απλά την εφαρμογή του άρθρου 7 όπως και για την Πολωνία. Βρισκόμαστε εδώ μάρτυρες μιας διαπιστωμένης παράβασης. Έχει υπάρξει απόπειρα παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Και υπάρχει πρόταση νόμου που καθιστά συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις μη τροποποιήσιμες εκ των υστέρων. Όλα αυτά νομίζω είναι επαρκή έτσι ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο 7 και αυτό ακριβώς προτείνουμε σε συνεργασία και με την Μπάρμπαρα Σπινέλη. Καλώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Τότε να ζητήσω παρακαλώ από τη Μαϊτέ να κλείσει τη συζήτηση σύντομα να ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία την οποία επέδειξαν. Θα συνεργαστούμε στενά και θα καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες να είναι ε, συνενετικές και λογικές. Ευχαριστώ. Να ζητήσω κάτι στα ισπανικά, λέει η κυρία Ούμπνα. Εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε στις 21 Μαρτίου ή στις 25 Απριλίου. Αν θέλεις λίγο χρόνο περισσότερο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε είτε στις 21 Μαρτίου είτε στις 25 Απριλίου. Προτιμάω τον Μάρτιο, λέει η κυρία Ρούις. Καλώς. Λοιπόν, η ψηφοφορία, επαναλαμβάνω, λέει η κυρία Χρύμπνερ, θα γίνει στις 21 Μαρτίου στην Επιτροπή μας. Να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού νόμου το 16. Εδώ είναι ο κύριος Βιεζόσκης ηγητής. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ήδη ήμουν εισηγητής μιας έκθεσης για την ε, υλοποίηση κάποιων νομοθετικών πλαισίων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση λοιπόν, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες και υπάρχει το γνωστό άρθρο που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μας ε, απασχολούν ιδιαίτερα οι κάποιες αρνητικές ε, διαδικασίες ε, του 2016. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι οι τάσεις δεν ήταν καθαρά θετικές, υπήρξαν πολλές παραβιάσεις, διαδικασίες, αναβολές, καθυστερήσεις για την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και αυτό σε πολλά κράτη και ε, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ε, τα πρότυπα για την καλύτερη νομοθεσία. Θέλω να αναφέρω εδώ και τη σημασία της διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντική η διαδικασία αυτή να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και όταν λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία αυτή αλλά και στην μεταφορά. Πιστεύω ότι πολλά σφάλματα μπορεί να αποφευχθούν με αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρώπη σήμερα αναρωτιούνται πού ακριβώς βασίζονται αυτές οι αποφάσεις. Και γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική και στην υλοποίηση και στην εφαρμογή και στη μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να παίρνει αποφάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους την ποιότητα και τη διαφάνεια. Αυτά είχα να πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις, σχόλια. Είμαι στη διάθεσή σας και βεβαίως θα ενσωματώσω τις στη γνωμοδότησή μου τις παρατηρήσεις σας. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του Ράινερ Βίλαν, που είναι ο σκιώδης εισηγητής εξ ονόματος της δικής μας πολιτικής ομάδας. Δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικό στην γνωμοδότηση αυτή λαμβάνονται υπόψη όλες οι προσφυγές, όλες οι περιπτώσεις παραβιάσεων που έλαβαν χώρα το 2016. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία που δεν λαμβάνονται υπόψη μου αρκετά ούτε από τη διαδικασία παρακολούθησης, ούτε από την γνωμοδότηση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι η ορθή μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται γλωσσική ακρίβεια, η σωστή ερμηνεία των λέξεων σε όλες τις γλώσσες, γιατί με μία λανθασμένη μετάφραση υπονομεύεται η ασφάλεια του νόμου. Χρειάζεται επίσης, ε, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο μου, η πολύ σοβαρή παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής και μεταφοράς του στην εθνική νομοθεσία και βλέπουμε ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πολλές φορές αναφέρουν αυτή την έλλειψη παρακολούθησης στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να πω ότι η κυρία Νταμπαρντέλη, η οποία είναι η συγγήτριά μας και η Όδης, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα. Μου έδωσε ένα μεγάλο έγγραφο εδώ, κείμενο, το οποίο θα δώσω στον εισηγητή. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα σημεία τα οποία θα έλεγα φέρνει στην επικαιρότητα το έγγραφό σας, στα γαλλικά θα τα πω, απαιτείται σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη να ξεκαθαρίσει ε, την κατάσταση και να βρει κάποιες λύσεις για, ε, ε, τα προβλήματα μεταφοράς, θα έλεγα, της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική. Νομίζω ότι είναι Πολύ συχνά τα προβλήματα αυτά της μεταφοράς θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε αν υπήρχε μια προληπτική βοήθεια για να γίνει η μεταφορά αυτή. Ε, μιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τα κράτη-μέλη σε τεχνικό επίπεδο σε σχέση με την διαδικασία επιπαραβάση, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις ε, οργανωτικές και θεσμικές τους ικανότητες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μειώσουν τις παραβάσεις Πάντως στόχος είναι αυτός τον οποίο είπα και όλα τα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να στηρίξουμε την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηριχθούν και να ενισχυθούν. Γι' αυτό και καταθέτω, όπως είπα, το έγγραφο αυτό στον συνάδελφο. Είναι στα γαλλικά, αλλά μπορώ να... εντάξει, το δέχεται στα γαλλικά λοιπόν. Θα σας το δώσω για να μην χάσουμε πολύ χρόνο τώρα. Σας ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος. Για τους πρασίνους δεν ξέρω. Για την FDD δεν υπάρχει κανείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση από πλευρά του εισηγητή. Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν, ευχαριστώ όλους που έκαναν παρατηρήσεις, ε, το κύριο Πρέντα, εκ μέρους του Σκιώδους. Σημείωσα όλα όσα είπατε, εκ μέρους ε, και των φιλελευθέρων και των σοσιαλιστών. Φυσικά και μπορώ να συμπληρώσω τη γνωμοδότησή μου με αυτά τα σημεία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην με βρίσκει σύμφωνο και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε παρατηρήσεις σε μια γνωμοδότηση και να την ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 2 Μαρτίου στις 12. Και κάτι που αντιτίθεται σε αυτό που είπε ο κύριος Βίλαντ, επειδή η ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι πολύ σύντομα, για να προλάβουμε θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν στα αγγλικά. Είπαμε λοιπόν προθεσμία υποβολής ε, των τροπολογιών 2 Μαρτίου, 21 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τις μεταφράσεις. Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική αν θέλουμε να προλάβουμε να υποβάλουμε τη γνωμοδότησή μας στην ε, τζούρι. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το θέμα της χρηματοδότησης των ε, πολιτικών ε, κομμάτων και ίδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμπαθάτε με γιατί η φωνή μου είναι χάλια, όπως βλέπετε, αλλά ελπίζω να τα καταφέρω με τη βοήθεια του μικροφόνου. Τώρα, συνολικά και γενικά, καλά πάνε τα πράγματα. Το Συμβούλιο συζήτησε τις προτάσεις μας. Και Όσοι από το πλήστον συμφωνήσανε, δέχτηκαν τις προτάσεις μας, τις τροποποιητικές, όμως διατυπώσανε κάποιες άλλες εναλλακτικέ προτάσεις σε τεχνικό επίπεδο ούτως ώστε να επιληθούν κάποια προβλήματα Α, και όλα αυτά εντάξει, απλώς τώρα έχουμε δύο θέματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν, πολιτικού χαρακτήρα. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την ισότητα των φύλων, μια που τα πολιτικά κόμματα τα οποία υπάγονται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ίδια τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα παρουσιάζουν στο website που έχουν τι, τι πρεσβεύουν σε πρώτη την ισότητα των φίλων σε σχέση ουσιαστικά με την προεκλογική εκστατεία για τις ευρωεκλογές Το δε συμβούλιο δεν μπορεί να σχετικά με αυτό και θέλει να φύγει η σχετική μνήμα. Δεύτερο θέμα που εκκρεμεί τώρα και ακόμα πιο αυστηρό όσον τη δική μας πρόταση. Είχαμε πει ότι θέλουμε να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την συνεχή δημοσιοποίηση του πολιτικού προγράμματος, του πολιτικού μανιφέστου, και του λογότυπου αυτών των ευρωπαϊκών ε, κομμάτων. Οπότε, αυτό το οποίο θέλει το Συμβούλιο είναι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν στα πολιτικά ευρωπαϊκά κόμματα να προσθέσουν το πρόγραμμά τους και το λογοτυπό τους ώστε να μπορέσουν να τύχουν χρηματοδότησης. Εμείς δε κατεβάσαμε το κατόφλι στο ελάχιστο 7. 7, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, γιατί δύο ο συνάδελφο ε, Βίλαντ ε, ανησυχούσε για το κατά πόσο να μπορέσουν όλα τα κόμματα να μπορέσουν να υπαχθούν, να τηρήσουν, να συμμορφωθούν προς αυτή τη διάταξη και Μιλάγαμε, ήρθαμε σε επαφή με τον συναδελφό Βίλαν για αυτή την ε, τροποποίηση, τροποποίηση του ΕΛΚ. Ούτως ώστε άμεσα να υπάρξει μόρφωση με αυτή την διάταξη. Να δούμε τώρα αυτά τα δύο σημεία, θα ζητούν στον τριμήρη διάλογο, αλλά θα εμείς να δούμε κατά πόσον τουλάχιστον εκουσίως να υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με την πολιτική της όντα των φίλων και από την άλλη μεριά να υπάρξει κάποια δέσμευση για το ζήτημα του αριθμού, για το ζήτημα του συνόλου των κομμάτων που θα πρέπει να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και το λογότυπο. Αυτά είναι τα δύο σημεία για τα οποία προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί συμφωνία εν ώψη του τριμερούς διαλόγου, ούτε καν σε επίπεδο τεχνικής συνάντησης πέραν των άλλων τροπολογιών και τροποποίησεων όπως σας προανέφερα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο τελικά να σημειωθεί αυτή η συμφωνία. Δεν στόχος είναι αύριο που έχουμε τη συνάντηση του τριμούς διαλόγου να τα βρούμε, οπότε το θέμα να κατέβει στην Ολομέλεια του Απριλίου, μια που πιέζει το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει αυτού του είδου η νομοθεσία, αυτό το καταστικό τέλο πάντων, να ισχύει όταν έρθει η ώρα των ε, εκλογών, όποτε και θα ενεργοποιηθεί και ο προπολογισμό. η πρικοδότηση για τις ε, εκλογές. Άρα ελπίζουμε να πετύχουμε το στόχο μας αύριο και έτσι να ολοκληρώσουμε να υπάρξει ένα συμβασμός λογικός. Ναι, δεν είναι και τόσο φοβερά αυτά τα δύο σημεία. Καλά, για, για μας είναι λίγο πιο περίπλοκο θέμα το ισότητα των δύο φίλων, αλλά λογικό. Μου φαίνεται μια από το Κοινοβούλιο συνεχώς πιέζει όσον αφορά ε, την πολιτική της ισότητας των φίλων. Ε, γι' αυτό και ζητούμε ότι τα πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουν χρηματοδότηση θα πρέπει να αναφέρουν, θα πρέπει να εκθέτουν στα website τα οποία διατηρούν το τι πολιτικές άγουν όσον αφορά αυτή την υπόθεση για τις υποψηφιότητες, για το προεκλογικό πρόγραμμα. Έτσι θα πρέπει. Και έτσι θα πρέπει να εμφανίζονται και οι γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Ε, τέλος πάντων, ελπίζω ότι τελικά θα τα βρούμε. Thank you very much, Mercedes, ε, for... Ευχαριστώ, Mercedes. Κύριος Μέσσερ για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στενά παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων και είμαι θα ικανοποιημένη με τη συμφωνία όσον αφορά το κατόφλι. Ε, από ό,τι κατάλαβα, μπορούμε να τα βρούμε και να ευχαριστήσουμε τους συγητάς. για την ευελιξία που έχουν επιδείξει. Προβληματίζομαι για κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί γιατί αυτά έχουν ανακύψει στα μέσα ενημέρωση, στις συζητήσεις σε με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα Πού είναι οι αλλαγές που επιφέρουμε. Τέλος πάντων, πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια. Και φαντάζομαι στο μέλλον θα συνεχίσουμε την ζήμωση για όλα αυτά. Τέλος πάντων, εάν τα πράγματα μείνουν έτσι, αν δεν αλλάξει τίποτα, σε σχέση με όσα συζητήσαμε ισχυώδης, ελπίζω ότι ο συμβασμός θα εξευρεθεί. Ή πρόεδρος, δεν βλέπω να υπάρχει εδώ πέρα συνάδελφος της ε, Άλντε Χέλμουτ Σόλτ δεν είναι εδώ. Το κύριο Σελίμοβιτ ούτε για το EFTD ούτε για το ENF. Α, έχετε το λόγο εσεί, κυρία Τζέιμ. Ναι, ναι, ναι, έχω ξαναθέσει το θέμα των πολιτικών κινημάτων και θα σα το ξαναπώ μια που έχουμε εξελίξει τι τελευταίε εβδομάδε στο Ηνωμένο Βασίλειο νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί Κάπου ε, γράψαμε εμείς ότι δεν θα γίνει το Brexit. Δεν είναι έτσι. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι στη Γαλλία έχουμε το όνομά το οποίο ήταν ένα κίνημα και όχι κόμμα. Το Ρινιό του Ηνωμένου Βασιλείου, του επεστήριξε ο Μακρόν και υπάρχουν και άλλες οργανώσεις διάφορα κρατημέλη τα οποία κινούνται σε αυτό το μήκος κύματος. Αφού έχουν έτσι τα πράγματα, στην έκθεσή μας το θίγουμε το ζήτημα. Εγώ δεν το νομίζω και γι' αυτό και σας το λέω. Γιατί εάν δεν γίνει το Brexit, ε, τότε θα συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές του 2019 και το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας θα είναι πολύ διαφορετικό. Θέλει κάποιο το λόγο, ίσω η Επιτροπή. Όχι, όχι, λέει διανεύματο. Κύριε Άνταμ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια από μέρους της Επιτροπής. Όπως είπαμε νωρίτερα, βεβαίως και θεωρούμε ότι ως έχει η σημερινή πρόταση μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιπτώσεις καταχρήσεων. Ο τριμερής διάλογος βέβαια έχει ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συζητείτε, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κάποια τεχνικά θέματα, όπως είπε και η συγγήτρια. Είμαστε διαθέσιμοι σε περίπτωση αν θέλετε, που θα χρειαστούν κάποιες διευκρινήσεις τεχνικές και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους, λέει η κυρία ότι ήδη έχουμε εξετάσει το κείμενο και το Συμβούλιο επίσης έχει ψηφίσει το κείμενο και βρισκόμαστε θα έλεγα στην τελική φάση στην ουσία συγκρίνουμε τα έγγραφά μας, προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι διαφορές πάνε στις οποίες μπορεί να υπάρξει μια κάποια συμφωνία. Ξέρω ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει και μόνο τα σημεία τα οποία συζητάμε σήμερα ε, είναι αυτά τα οποία είναι αντικείμενο συζήτησης. Μιλάμε για πολιτικά κόμματα καταγεγραμμένα που σέβονται δηλαδή το σύνολο της διαδικασίας όπως προβλέπεται για την καταγραφή, κινήματα και κόμματα τα οποία προβλέπεται ο κανονισμός λειτουργίας τους από τον νόμο, αν κάποιος θέλει να καταγραφεί σαν πολιτικό κόμμα και να έχει την δυνατότητα σε οικονομική βοήθεια θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες και σε αυτή την περίπτωση οι κανόνες αλλάζουν στην περίπτωση αυτή σε σχέση με την ενημέρωση η οποία δίδεται προς το κοινό και στις εγγυήσει για να μην υπάρξει κατάχρηση σε σχέση με το δημόσιο χρήμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως σε σχέση με την πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις αυτές εφόσον δεν γίνονται σεβαστοί οι όροι. Και εδώ μπορεί να υπάρξει παραπομπή επίσης και αναφορά στον, στην οδηγία η οποία ρυθμίζει την λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Πάντως, τα σημεία τα οποία έχουν τεθεί σε συζήτηση είναι αυτά στα οποία υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο. Είναι λίγα τα σημεία αυτά, δύο βασικά, και τα υπόλοιπα είναι θα έλεγα κάποιες μικρότερες δυσκολίες τις οποίες θα βρούμε εύκολα μια λύση. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι στο μέλλον θα επανέλθουμε στο θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων σε μεγαλύτερο βάθος Πάντως επαναλαμβάνω ότι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο για την Επιτροπή, ξαναλέει ο ομιλήτρια. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκουμε να πετύχουμε, αλλά δεν το βρίσκω σημαντικό και θα βρεθεί λύση εύκολα. Thank you very much, ε, Ευχαριστώ τη Μεσέντες. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αύριο στην τεχνική συνάντηση θα διευκρινίσουμε τις εναπομείνασες διαφορές και στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου θα βρούμε την τελική λύση. Το Προεδρείο θα πρέπει να εφαρμόσει τις εφαρμοστικές, να εγκρίνει τις εφαρμοστικές διατάξεις και την εφαρμογή του στον προϋπολογισμό του 19 πριν το τέλος Ιουνίου δηλαδή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τελικά στις αρχές Μαΐου το αργότερο. Και αν είναι δυνατόν και νωρίτερα, λέει η κυρία Μπρέσο αλλά θα είμαστε ευέλικτοι και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε την διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, να τελειώσουμε με το θέμα αυτό. Ο κύριος Σόπλιν δεν χάθηκε. Οπότε θα έχουμε ένα διάλειμμα. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν στις, 10, 5 και 15. Ελπίζω να βρεθούμε όμως στις 5, μην τυχόν και έχει επιστρέψει μέχρι τότε ο κύριος Σέπλιν. 5 παρακαλώ να είστε πίσω στις 5. Έχετε ε, αρκετή ώρα μέχρι τις 5. Thank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

Ευχαριστώ.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

Πάντω.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

Colleagues, we still have one minute. Maybe we check the cards in the meantime. Because... Η Πρόεδρος, ας ψηφίσουμε γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οπότε να βάλετε την κάρτα παρακαλώ στην συσκευή ηλεκτρονική ψηφοφορία να κάνουμε δοκιμή. You Is abstaining a vote cast? Αποχή, ψηφίσατε όλοι η Paradigma Παραδείγματος χάρη τονίζει πρώτα. Okay, 19, 18, voting, no, 20, 19. Okay, more or less. Let's see the result. Okay. Really adopted. Okay, I think it's Okay. No, it's 14. I was once criticized for starting too early. <laughs> Μήπως δεν ήρθε η ώρα ακόμα, λέει η πρόεδρος, και κοιτάει το ρολόι που λέει ένα λεπτό νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα. Α, δεν είναι εδώ η συνάδελφος. Τέλος πάντων, τότε να αρχίσουμε. Αλλά πρώτα, μην ξεχνάτε συνάδελφοι, ότι έχουμε δύο εκθέσεις. Είναι της Mercedes και του Καστάλτο. Πρόκειται για υπηρεσίες και για την έκθεση αυτήν δεν τα συζητήσαμε. Άρα για την υπηρεσία φαρμάκων ας δώσουν πρώτο λόγο στην Mercedes. Συνάδελφοι, γνωρίζετε πώς πήγαν τα πράγματα. Σημειώθηκε διοργανική συμφωνία η οποία καθόριζε το πλαίσιο αποφάσεως όσον αφορά την έδρα αυτής της υπηρεσίας. Και συζητήθηκε ο ρόλος των συνομοθετών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Προχώρησε η διαδικασία με οίκιστα διαφανή τρόπο δεν υπήρξε ενημέρωση προς τους συνομοθέτες και συγκεκριμένα προς το Κοινοβούλιο. Δεν έκανε κανείς συμφωνητή στο το Συμβούλιο. Το έκαναν τα μέλη αυτού. Οι 27 πλην Μεγάλης Βρετανίας. Και συνήφθη η συμφωνία και επικυρώθηκε με μία ε, κλήρωση. Ούτε καν πρακτικά δεν έχουμε. Τι συζητήσουμε, αγνώμε τα πάντα, δεν ξέρουμε τι έγινε, πώς. Τι, τίποτα δεν ξέρουμε. Το Κοινοβούλιο προέβησε σειρά δηλώσεων, κυρίως των ηγετών των πολιτικών ομάδων και κυρίως του Προέδρου. Και είπε ότι έτσι παραβιάζονται, παραβιάζονται το, το, το, το, πλαίσιο των νομοδιοτήτων, των νομοθετικών, παρά το ότι έπρεπε να ψηφίσει το κείμενο και επομένω ε, ανετράπει η συμφωνία που υπήρχε, άρα αναστέλλεται και ματαιών του για το μέλλον. Αυτά από τις ε, δηλώσεις και εμείς δεν έχουμε φαστηρική αρμοδιότητα, απλώς γνωμοδοτική δεν έχουμε την καθήλυν κυρίως αρμοδιότητα. Τέλος πάντων, το περίπου τα λέμε και εγώ και ο Καστάλτο. Και τονίζουμε το ότι χρειάζεται να γίνει άμεσα αναθεώρηση αυτού του common approach όπως αυτό έλαβε σάρκα και ως τα και λέμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να εμπλέκεται πολύ περισσότερο το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης της απόφασης ε, με δεδομένη την συνομοθετική του αρμοδιότητα. Και δεύτερον, είπαμε με κάποια δήλωση πώς έχουν αυτές οι βασικές αρχές και λέμε σε αυτή τη δήλωση ότι τα κριτήρια της επιλογής ε, δεν ε, στάθηκαν ικανοποιητικά και ότι καταδικάζουμε το ότι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με αυτού του είδους τον, τον, τον τρόπο αυτή την κλήρωση ούτως με μια διαδικασία καθόλου διάφανη και διαφανή. Και είπαμε ότι όλα αυτά θα πρέπει άρτη να αλλάξουν για το μέλλον. Επίσης έχουμε κάποιες τροπολογίες και τις υποφαινόμενες που τροποποιήθηκε από προφορική τροπολογία του συναδελφού Μπρόκ με τον οποίο συμφωνήσαμε. Και σε αυτή την τροπολογία αποσκοπούμε να ματαιωθεί η επιλογή που έγινε μέσα από αυτήν την ε, αδιάφωνη διαδικασία ε, παραβάση της διοργανικής ε, συμφωνίας του Άμστερνταμ. Και ότι αντί όλων αυτών θα πρέπει να σημειωθεί συμφωνία των συνομοθετών. Άρα να επανέλθουμε στη διαδικασία της συμφωνίας των δύο συνομοθετών. Οπότε, έτσι ήταν πιο αποφασιστική η διατύπωση σε σχέση με την διεκδίκηση υπέρ των αρμοδίων του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για κάποια διαμαρτυρία, αλλά τελικά εκυρώσαμε τη σχετική απόφαση. Και δυστυχώ τα πράγματα πάρα πολύ συχνά γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Με δυσκολία απόφαση και όπως είπαμε πρόκειται για γνωμοδότηση δική μας προς την ένβη. Και ευτυχώς χαιρετίζουμε το γεγονό το ότι το Κοινοβούλιο όχι δια της Επιτροπής μας λαμβάνει υπόψη το έγινε, προσέχει τις αρμοδιότητές μας αλλά από την άλλη μεριά δεν αποτελεί διεκδίκηση το ότι επικυρώσαμε την σα συμφωνία και πάλι συμφωνώ, ε, για τη φωνή. Συνάδελφοι, τώρα να ακούσουμε και τον Φάμπιο, αλλά δεν ήρθε. Θέλει κάποιος να μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Καστάλτο. Α, εσείς. Ένα θέλω να πω. να επαναλάβω ότι οι δύο γνωμοδοτήσεις είναι παρόμοιες και ότι και στη γνωμοδότηση του Καστάλτο Στόχος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει ε, ό,τι δυνατό και να εφαρμόσει όλες τις αρμοδιότητες της, να ασκήσει μάλλον όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται. Καλώ σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Α, ο Άντερσον. Ευχαριστώ. Δεν είναι δικό μου βέβαια το θέμα αυτό, αλλά κατάλαβα καλά αυτό που λέει η κυρία Μπέζο. Θέλει να ψηφίσουμε ουσιαστικά κάνοντας μία σύσταση προς την ένβη με τον κίνδυνο αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα να μην ουσιαστικά προλάβουμε να πάρουμε την απόφαση γέρος για τον Brexit. Κατάλαβα καλά. Ο κύριος Κόρμπετ προτείνει να καθυστερήσουμε τον Brexit. Καταλαβαίνω ότι σκέφτεται, αλλά τώρα ας είμαστε λίγο σοβαροί. Το να καθυστερήσουμε την απόφαση όσον αφορά το πού θα μπει η έδρα αυτού του οργανισμού. Δεν νομίζω ότι θα, καθυ... θα καθυστερήσει καθόλου το Brexit. Τι προτείνουν οι εισηγητές, κατάλαβα καλά την πρόταση των εισηγητών. no, no uh, intervention. Δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν ξέρω, δεν, δεν θέλω να πάρω το λόγο, ίσως να ήταν κάποιοι άλλοι που ήθελαν το λόγο πριν, επιβεβαιώνω το ότι υπάρχουν δύο τύποι προτάσεων. Η πρώτη έχει σαν στόχο στα πλαίσια του νομοθετικού, ε, της νομοθετικής πρότασης να επαναλάβουμε με μία ξεχωριστή δήλωση τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δεύτερη πρόταση είναι η προφορική τροπολογία στην τροπολογία 8 στα πλαίσια της τροπολογίας προφορικής να βγάλουμε τη λέξη Άμστερνταμ, την επιλογή Άμστερνταμ και να βάλουμε μια συμπεφωνημένη λύση ανάμεσα στους δύο συνεισηγητές. Εφόσον βρείτε ακριβώς την τροπολογία 8. Λέγεται εκεί ότι θα πρέπει να ακολουθεί η τακτική νομοθετική διαδικασία υπενθυμίζοντας ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτες και θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές και προσωρινές εγκαταστάσεις. Γιατί ξέρετε ότι υπήρξαν κάποιες νέες μορφές ενημέρωσης και από ό,τι φαίνεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη γιατί όπως πάρα πολύ συχνά η προσπάθεια την οποία έκανε το Συμβούλιο, δεν ήταν καν το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο έτσι κι δεν έχει ψηφίσει ακόμα, ήταν η ε, απλή συνάντηση των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ιδιαίτερα σκοτεινή, και ε, επί τη βάση των πληροφοριών ε, οι οποίες δόθηκαν και οι οποίες εν πολλής απεκρίβησαν δεν μας οδηγούν στο να δεχθούμε απόλυτα την πρόταση. Το Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση αγνοήθηκε πλήρως από όλη την διαδικασία παρότι είναι συνεισηγητής και κανονικά ο συνεισηγητής θα πρέπει να είναι πάντα ενήμερος της διαδικασίας και ενήμερος των πληροφοριών που πηγαίνουν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Θέλει κάποιος άλλες εξηγήσεις γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, είναι σαφές, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα, θα ψηφίσουμε για την εξωτερική υπηρεσία φαρμάκων. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 8. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Μιλάω για την προφορική τροπολογία. Δεν ψηφίζουμε την 8. Ρωτώ αν κάποιος είναι κατά της προφορικής. Κανείς δεν είναι κατά. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 8 τροπολογημένη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote is closed. And it is rejected. It looked close, but it's strongly rejected. 7 to 14 to 1. So we go to... Λοιπόν, 14 κατά, 7 υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 6. Φάμπιο Καστάλντο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση βέβαια εκ των υστέρων. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η σωστή θέση για την συγκεκριμένη αυτή αναφορά. Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο νομικά το θέμα. Ε, θα ψηφίσουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χάσουμε. Ποιοι είναι υπέρ της 6. Κατά. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 6. Ψηφίζεται. Τέλος δεκτή. 12 υπέρ, 10 κατά. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 7. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορία. Απερίφε. Τώρα περνάμε στην προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος και για την προφορική ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίας. Δεκτή. 14 υπέρ 8 κατά. Περνάμε τώρα ε, στο σύνολο του... Α, όχι, για μια στιγμή. Ναι, το σύνολο του ψηφίσματος. Διακόπτει η πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. 12 υπέρ 10 κατά. Συμβιβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι, λάθος λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 3. Διακόπτη πάλι η πρόεδρος. Διακόπτη η πρόεδρος. Λοιπόν, συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τώρα έρχεται η τελική ψήφος. Ονομαστική κλίση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος δεν ψηφίζει. Α, όχι, όλοι ψήφισαν. Λοιπόν, 18 υπέρ, 3 κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην νομοδότηση Καστάλτο. Ε, για την τροπολογία 5 υπάρχει η αμφιβολία ότι μπορεί να τεθεί ένα πρόβλημα σε σχέση με τη νομική βάση. Δεν ξέρω ποιος θα το εξετάσει. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε για το σύνολο της νομοθετικής πράξης. Ψηφίζεται. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. Τώρα, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη. Οπότε ψηφίζουμε για την τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα, ονομαστική κλίση για το σύνολο της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 3 κατά, δεκτό. Περνάμε τώρα. Στην έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Ψηφίζετε παρακαλώ. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά ποιος θα το πει. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 7 υπέρ 15 κατά. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. αλλάζετε τη γνώμη σας, ως εκ τούτου θα πρέπει να ελέγξουμε την 10. Ψηφίζετε για την 10. Ηλεκτρονική ψήφος για την 10. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 όχι όχι 20 λάθος 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική β υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Β παρακαλώ ψηφίζετε. Πέραση της ψηφοφορίας. 15 υπέρ 7 κατά δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 23 δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ, 34 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 36 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 37. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη εκ νέου. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 39 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη, 40 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 41 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Ονομαστική κλίση για το σύνολο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 21 υπέρ, ένας κατά. Δυστυχώς χάσαμε τον κύριο Σέπλιν. Οπότε δεν μπορούμε να τον περιμένουμε. Δεν έχετε κανένα νέο από τον κύριο Σέπλιν. Όχι. Καλώς λοιπόν, τέλος της συνεδρίασης θα προσπαθήσουμε να βολέψουμε τη συζήτηση Σέπλιν αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.